Παρακαλώ, ο κύριο Σαλάτο. Με συγχωρείτε, Πρόεδρε. Θα παρακαλούσα η πρόεδρο Κρόπερκ να είχε παρέμβει και σε παρόμοιες ε, περιπτώσεις για να έχουν απελευθερωθεί και πολιτικό κρατημόνιο στο Ιράκ, πέρα από αυτό που είπε σήμερα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και η κυρία Σουίκα. Η κυρία Σουίκα δεν είναι στην αίθουσα. Μία ανακοίνωση τώρα. Βάσει του άρθρου 216 εδάφιο 4 σας ενημερώνω ότι δεν υπάρχει καμία αίτηση για να εφαρμοστεί στις ψηφοφορίες στο διευθυντικό που ανακοινώθηκε.